Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να χαιρετήσω για άλλη μια φορά την πολύ καλή αυτή πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Δαμανάκη. Ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημέρα διάταξη είναι η έκθεση Σαλαβράκου περιορισμή στην Αλία και στα χωρικά ύδατα Μεσογείου και Μαύρης θάλασσα και δίνω αμέσως το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδέλφοι, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν πάνω στη συγκεκριμένη έκθεση και χάρη στην καλή συνεργασία που είχαμε καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε ένα συνεκτικό κείμενο που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Αλίας μεγάλο τμήμα της θαλάσσιας επιφάνειας της μεσογείου βρίσκεται σήμερα εκτός της δικαιοδοσίας ή της κυριαρχίας των παράκτιων κρατών. συνεπώς παραμένει σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτο όσον αφορά τους έμβιους υδρόβιους πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον τους. στην έκθεσή μου γίνεται προσπάθεια απεικόνησης του προβλήματος και διατυπώνονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις αλλιευτικές ζώνες και τη διαχείριση της ελίας. Γίνεται ξεκάθαρο φυσικά ότι βάση είναι η υπάρχουσα νομοθεσία των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διεθνές δίκαιο και κυρίως η σύμβαση του ΟΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας η Ανκλός. Από τα 21 μεσογειακά κράτη μόνο τρία δεν έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση του ΟΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Πρόκειται για το Ισραήλ, τη Συρία και την Τουρκία. Δεδομένου όπως προελέχθη ότι η σύμβαση αυτή είναι μέρος του διεθνούς δικαίου για τη διαχείριση των υδάτων και των αλλιευτικών πόρων θα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να χρησιμοποιήσει τα διπλωματικά της μέσα ώστε οι χώρες αυτές να υπογράψουν τη σύμβαση και ειδικότερα οι χώρες που βρίσκονται υπό ενταξιακό καθεστώς. Η θαλάσσια διαχείριση, η προστασία του θαλασσιού περιβάλλοντος και των αλλιευτικών πόρων καθώς και ο έλεγχος για την παράνομη άναρχη και λαθρέα αλληλεία έχει αποδειχθεί ότι προστατεύεται καλύτερα όταν υπάρχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο. κατά αυτόν τον τρόπο μέσα από την έκθεσή μου ενθαρρύνεται η δημιουργία θαλασσίων ζωνών και ειδικότερα η ανακήρυξη αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και καλείται η επιτροπή να συνδράμει στον τομέα αυτό παρέχοντας ανάλογη καθοδήγηση στα κράτη μέλη. τονίζεται βεβαίως ότι αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητος η δημιουργία και ο καθορισμός του ΩΣ είναι αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών που θα σταθμίσουν τα δικά τους συμφέροντα εν προκειμένου και θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. ευχαριστώ την κυρία επίτροπο για την παρέμβασή της και χαιρετίζω τις προσπάθειες της επιτροπής ε, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στα πλαίσια της στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη καθώς και την πρόσφατη μελέτη της επιτροπής που εξετάζει το κόστος και το ωφέλη της θέσπισης των θαλασσίων ζωνών στη μεσόγειο και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες θα είχε θετικά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές της γαλάζιας ανάπτυξης προσελκύοντας επενδύσεις και περαιτέρω οικονομικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Nous Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία Καστιάη. Ο κύριος Στίερ έχει το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία του εισηγητή και να υπογραμμίσω δύο στοιχεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Πρώτον όσον αφορά το σεβασμό του διεθνούς δικαίου όταν πρόκειται για διαμάχες όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 του σχέδιου ψηφίσματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να ισχύσει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Θαλάσσιο Δίκαιο. Πιστεύω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η σύμβαση του 61 να ισχύσει εδώ βασιζόμενη πάντα σε κριτήρια δικαίου και όχι πολιτικά. Και εδώ αναφέρομαι στη μάχη μεταξύ κρατίας και Σλοβενίας. Το άρθρο 15 επίσης είναι πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρεται στις ΑΟΣ. θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και υπενθυμίζω ότι η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου μπορεί να επιτρέψει εδώ να προστατεύσουμε την Μεσόγειο. Hvala ο κύριος Πίγουλα, ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής αναφέρεται στις διάφορες συναλλαγές παράνομες οι οποίες πολλές φορές κινδυνεύουν να καταστρέψουν κάποιες θαλάσσιες περιοχές. Στη Μεσόγειο τα προβλήματα είναι τέτοια που χρειάζεται μια ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεράσουμε διαμάχες στην Αδριατική, παραδείγματο χάρη, η διαχείριση των αλλιευμάτων μεταξύ των διαφορετικών στόλων, θα πρέπει να διέπονται από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι παράκτιες περιοχές, νησιωτικές περιοχές σήμερα γνωρίζουν μείωση του πληθυσμού τους και απερίμωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ στην περιοχή της Κροατίας παραδείγματος χάρη να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε ότι η αλία έχει και μια πολύ σημαντική οικονομική συνέπεια για τους ε, εγχώριους πληθυσμούς. Και εγώ προέρχομαι από την ε, Κροατία, η οποία Βρέχεται από τις ε, δαλματικές ακτές και ξέρετε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει από την αλία. Γι' αυτό η προστασία της αλίας είναι ύψης της σημασίας. Χαίρομαι για το ψήφισμα αυτό που δεν θα επιτρέψει την υπεραλίευση και την υπερεκμετάλλευση των αλλιευτικών χώρων. Μέσα στα πλαίσια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κάθε χώρα θα μπορέσει να προστατεύσει τους αλλιευτικούς της πόρους. Έτσι θα μπορέσουμε να ε, μειώσουμε αυτή την υπεραλίευση και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μακροπρόθεσμα. Καλό την Επιτροπή να λάβει θέση επί του θέματος και να μας προτείνει απτά μέτρα μέσα στα πλαίσια αυτού του ψηφίσματος. Η κυρία Σουίτσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Ξέρουμε ότι η Ελία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας που δημιουργεί πολλές θέσεις απασχόλησης και από την άλλη παρέχει πάρα πολλά τρόφιμα για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Έχουμε όμως και κάποια φαινόμενα υπεραλίευσης στην Μεσόγειο και ιδίω στην Αδριατική θάλασσα, περιοχή από την οποία προέρχομαι. Η υπεραλίευση πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τη βιώσιμη χρηστή διαχείριση της αλίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτήων ζωνών. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα πλέον για την Μεσόγειο, στα πλαίσια του οποίου θα μας σε να προστατεύσουμε τους ελευτικούς πόρους και επομένω στηρίζω πλήρω την προσέγγιση που προβλέπεται στην έκθεση. Ευχαριστώ κύριο Μίλαν. Να συγχαρώ τον κύριο Σαλαβράκο για την εξαιρετική εργασία. Κύριε Πίτροπε, το θέμα είναι πολύ απλό. Τι σημαίνει η έκθεση πρωτοβουλίας. Όταν διανοίγουμε μία δόση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιμένουμε από την Επιτροπή συγκεκριμένες δράσεις. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω μία προσέγγιση στην έκθεση πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι εμπεριέχει η Μεσόγειος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν επέλθει πολλοί κλειδονισμοί στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό η ευρωπαϊκή μας πολιτική αλληλείας θα πρέπει να ορίζει την συμπεριφορά των κρατών μελών στη θάλασσα αυτή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, ε, έχουμε και 14 χώρες που δεν είναι ευρωπαϊκές. 8 είναι ευρωπαϊκές, 14 όχι. Και αυτό δεν επισυμβαίνει πέρα από συγκεκριμένες διεθνείς συμφωνίες. Θα πρέπει λοιπόν να αποτανθούμε σε αυτές τις χώρες με συμφωνίες. Συζητήσαμε την αλλιευτική συμφωνία με τη Μαυρο... Μαυριτανία το απόγευμα. Δηλαδή πρόκειται για μια συμφωνία για το πώς θα γίνει η αλλίευση στα ύδατα της Μαυριτανίας. Γι' αυτό θα πρέπει να συνάψουμε αλλιευτικές συμφωνίες στη Μεσόγειο χωρίς το αντικείμενο να είναι η αλίευση κάθε αυτή, αλλά η τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων από όλους. Εάν από την έκθεση του κυρίου Σαλαβράκου ε, απορρεύσει μια τέτοια πρωτοβουλία, τότε θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την αλία. Ευχαριστώ την Πρόεδρο που ήταν ανεκτική ως προς το χρόνο παρέμβασης αλλά είναι και η τελευταία μας έκθεση. Ακριβώς και γι' αυτό έγινε και αυτή η εξαίρεση και δίνω το λόγο στην Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Και εγώ χαιρετίζω την έκθεση του κυρίου Σαλαβράκου. Συμφωνώ με την γενική του ανάλυση όσον αφορά την κατάσταση. Βεβαίως, η θάλασσα αποτελεί πηγή οικονομικής ανάπτυξης και φυσικά και θα πρέπει να είναι βιώσιμη η διαχείριση των ε, αληθικών πόρων. Μας χρειάζεται ένα πλαίσιο ισχυρό, ένα καλό σύστημα διακυβέρνησης, μια καλή και χρηστή διαχείριση των πόρων, έλεγχος και φυσικά η ενίσχυση και η εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται περιφερειακά. Αυτό ισχύει και για τη Μεσόγειο και για τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί χρειάζεται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό συντονισμένο επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε αυτά που αποφασίσαμε και να ενισχύσουμε τις νομοθεσίες μας είτε ε, πρόκειται για τους ολιεκτικούς πόρους είτε πρόκειται για το περιβάλλον. Συμφωνώ όμως κύριε Μιλάνα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε και τις τρίτες χώρες, τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμφωνήσουν, να συμβαδίσουν μαζί μας έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τις συγκρούσεις είτε να βρούμε έναν ε, ομαλό διακανονισμό, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Οι περισσότερες παράκτιες χώρες και στην Μεσόγειο αλλά και στην Μαύρη Θάλασσα δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως η ζώνες αποκλειστικής ε, οικονομικής εκμετάλλευσης δεν ανήκουν ε, αποκλειστικά στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται στρατηγικός διάλογος και πρωτοβουλίες για την ε, διαρρύθμιση των διαφορών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ακολουθήσουμε και βεβαίως η GFCM αλλά και η διευθέτηση των αλλιευμάτων του Ατλαντικού, του τόνου παραδείγματος χάρη, οι επιτροπές αυτές και οι πρωτοβουλίες αυτές, καθώς και άλλες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οδηγήσουν στην αναθεώρηση αυτών των συμφωνιών. Χρειαζόμαστε καλύτερα στοιχεία, καλύτερη συλλογή στοιχείων, βασιζόμενη σε επιστημονικά δεδομένα και μηχανισμούς και σχέδια τη διαχείριση των πόρων έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την παράνομη και λαθρέα αλία, άναρχη και λαθρέα αλία. Η Τουρκία, η Ρωσία, η Ουκρανία θα πρέπει να συμβαδίσουν μαζί μας, να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια για διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της αιματοφύλακα των συνθήκων και συντονιστή αυτής της πολιτικής, αλλά και τα κράτη-μέλη και οι εταίροι μας τρίτες χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν την εκμετάλλευση με χρηστό βιώσιμο τρόπο σε συνεργασία με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ασχίσουν οι πρωτοβουλίες για την Αδριατική, το Ιόνιο και τη Μαύρη θάλασσα. Η θέσπιση ΑΟΣ βεβαίως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κάτι που προϋποθέτει την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ε, τρίτων χωρών για να υπάρξει συντονισμός και υιοθέτηση, εφαρμογή των ε, μέτρων που έχουν ληφθεί. Μια πρόσφατη μελέτη μας οδήγησε στην πρωτοβουλία για περισσότερη συνεργασία στη Μεσόγειο με σκοπό όλες οι παράκτιες χώρες να μπορέσουν να ε, λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως είμαστε πολύ θετικά διατεθειμένοι προς αυτό. Μάλιστα, επεξεργαζόμαστε μία πιθανή πρωτοβουλία έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα δικαιώματά τους στο καθεστώς της θέσπισης ΑΟΣ για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη της γαλάζιας και την πρόθεση της γαλάζιας ανάπτυξης. Ολοκληρώνοντας, θα πω αυτή την εξαιρετική έκθεση και την αναγνώριση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν πιο ισχυρό και διαρθρωμένο διάλογο με τις τρίτες χώρες. Θα ήθελα εδώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, η χρηστή εκμετάλλευση των πόρων και η καλύτερη συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Θα συνεδριάσουμε αύριο 8 Οκτωβρίου από τις 8.30 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 19 ε, μέχρι τις 7 το βράδυ λύεται η συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.